Allow me to declare the meeting open. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Πολιτισμού. Ονομάζομαι Πάουλ Σμιτ και ήμουν πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται απευθείας. Στόχος μας είναι οι αρχαιρεσίες του Πρόεδρου και των Αντιπρόεδρων συγκεκριμένα, των τεσσάρων Αντιπρόεδρων, με βάση το, κανόν, το άρθρο 191 του εσωτερικού κανονισμού. Καταρχήν θα πρέπει να εκλέξουμε τον Πρόεδρό μας και μετά διαδοχικά τους τέσσερις Αντιπρόεδρους μας. Σημείο 2 της διάταξης, εκλογή του νέου Πρόεδρου της Επιτροπής Πολιτισμού. πρώτα απ' όλα να εξακριβώσουμε την απαρτία μας. Ένα τέταρτο των παρόντων μελών. Επειδή δεν σας γνωρίζω προσωπικά, θα μπορούσατε να σηκώσετε το χέρι σας αν είστε τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής. Παρακαλώ για να εξακριβώσουμε την απαρτία. We have the quorum. Yes. Uh, now I ask for nomination. Καλώς υπάρχει απαρτία. Τώρα υποψηφιότητες για τη θέση του Πρόεδρου. Yes, please. Could you tell your name, please? Because... Μάρκος Κούρια. Μάρκος Κούρια λέγομαι. Προτείνω πρόεδρο την κυρία Πακ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Is there any other nomination? Άλλες υποψηφιότητες για τη θέση αυτή. Αν όχι, μια και έχουμε έναν υποψήφιο, Νομίζω ότι μπορούμε να εκλέξουμε διαβοή στην κυρία Πακ. Συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Πακ και σας καλώ να πάρετε τη θέση του Προέδρου. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και στα αγγλικά μετά από τα γερμανικά. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί στην Επιτροπή ε, Πολιτισμού τόσους πολλούς και τόσο γεμάτη αίθουσα, σας το λέω αυτό. Χαίρομαι που μου δώσατε την εμπιστοσύνη σας. 20 χρόνια εργάζομαι στην Επιτροπή Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επί 17 έτη Ήμουν συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και τώρα δυσκολεύομαι κάπως να βγω από το πετσί της συντονίστριας και να ανέλθω σε αυτά τα ύψη του Προεδρείου, όπου θα πρέπει πάντα να είναι κανείς υπερκομματικός. Αλλά θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Γιατί εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού, ανέκαθεν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία. Και στην πολιτισμένη συμβίωση και συνεργασία προσβλέπουμε. Ερχόμαστε λοιπόν στο σημείο 2 τώρα της ημέρης της δέταξης. Στο σημείο C3 που είναι η εκλογή του πρώτου αντιπρόεδρου. Η εκλογή του πρώτου αντιπρόεδρου. Η απαρτία έχει ήδη διαπιστωθεί, είναι δεδομένη και έχουμε μία υποψηφιότητα, μία συνάδελφο, παρακαλώ να προτείνετε ε, την κυρία αυτή. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας συγχαίρω για την ε, πρόσφατη εκλογή σας. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα από την ομάδα των Πρασίνων την, να προτείνω την Έλκε Τρούπελ για την θέση της πρώτης Αντιπροέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού. Η Έλντα τα πέντε προηγούμενα χρόνια έδειξε την δέσμευσή της για να ε, προωθήσει την ε, πολύμορφη Ευρώπη και το διαπολιτιστικό διάλογο. Έδειξε επίσης ε, ότι η Ευρώπη πιο κοντά στον πολίτη, μια Ευρώπη της γνώσης είναι πολύ σημαντική. Ασχολήθηκε με τον οπτικοακουστικό τομέα και με τα δημοσιονομικά θέματα. Ζητώ εκ μέρου τη ε, συγγνώμη σήμερα. Έχει ανηλυμένε υποχρεώσει και δεν μπόρεσε να έρθει. Αλλά θα συνεχίσει τι προσπάθειές τη και πιστεύω, πιστεύω και εγώ και οι πράσινοι ότι θα είναι θαυμάσια αντιπρόεδρο για την Επιτροπή του Πολιτισμού και τη Εκπαίδευση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω το εξή. Υποσχέθηκα στη Χέλγα Τρούπελ ότι ε, θα σας, σας εξηγήσω γιατί η κόρη της ήταν σε ένα νησί στην Ελλάδα με τον πατέρα της και ασθένησε. Και τώρα ε, γύρισε πίσω και θα πρέπει να την πάει στο νοσοκομείο. Και πραγματικά έχουμε όλη κατανόηση γι' αυτό. Θέλω να ε, υπογραμμίσω αυτό που είπε η συνάδελφός μας. Η Χέλγα Τρίπελ τα τελευταία χρόνια δούλεψε πάρα πολύ καλά με όλους μας, συνεργάστηκε θαυμάσια και θα χαιρόμουν αν ψηφίζατε τη Χέλγα Τρίπελ. Υπάρχει άλλη πρόταση? Όχι διαβοή σας παρακαλώ να επιβεβαιώσουμε την εκλογή της. Ευχαριστώ πολύ. Και ερχόμαστε τώρα στην εκλογή του Δευτέρου Αντιπροέδρου. Εκόμα έχουμε απαρτία. Σας ερωτώ ποιος προτείνει ποιον. Κύριε Τάνου Τάκουλα. Ευχαριστώ. Σας συγχαίρω κυρία Πρόεδρε για την εκλογή σας. Θα ήθελα να αναφέρω τον Τίμο Σοίνη, ένα Φιλανδό βουλευτή, και να τον προτείνω ε, ο, για τη θέση του Αντιπροέδρου. Έχω δουλέψει στο Φινλανδικό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του, του Φινλανδικού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι πολύ επικοδομητική αυτή η πρόταση, γιατί είναι ε, διατεθειμένος να συνεργαστεί με όλους σας. Μάλιστα. Προτείνεται λοιπόν ο συνάδελφος κύριος Σόινη. Ε, άλλες αντιπροτάσεις έχουμε και αντιποψηφιότητες. Όχι, από το βλέπω. Η ε, κυρία Μπαντία, παρακαλώ. Sí, gracias, señora presidenta. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να ψηφίσουμε, όχι διαβοής, ε, τον αντιπρόεδρο αυτό, τον υποψήφιο αυτό. Μαρία, πείτε spe Εξ ονόματος των σοσιαλιστών, έχω ένα αίτημα για μυστική ψηφοφορία. Σωστά σας κατάλαβα. Θέλετε με σηκώνοντα το χέρι. Ναι, ναι, ναι, όχι μυστική ψηφοφορία, όπως να είναι. Θέλει κανεί μυστική ψηφοφορία. Όχι. Τότε, ποιο είναι υπέρ της εκλογής του κυρίου Σόινη. Δεν επιτρέπεται. Το φαντάστηκα, αλλά νόμιζα δεν θα το πάρει κανεί η ειδησία, αλλά το πήρε. Λοιπόν, Μαρία, τώρα μας επιφυλάσσει μυστική ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Παρακαλώ τη γραμματεία να μοιράσει χαρτιά, ψηφοδέλτια δηλαδή και παρακαλώ ε, να ορίσουμε και δύο ψηφολέκτες. Τι να κάνω, να σας τραβήξω κλήρο, όποιον δω. Μια που κάνουμε μυστική ψηφοφορία θα παρακαλούσα τον κύριο Σόινι τουλάχιστον να συστηθεί, αν μη τι άλλο. Mr. could Θέλετε να πάρετε το λόγο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Υπήρξε για 12 χρόνια πρόεδρος του κόμματός μου και μέλος της Φιλανδικής Βουλής για δύο συναπτές κοινοβουλευτικέ θητείες. Ήμουν στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, συμμετείχα και στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση και ασχολήθηκα με θέματα εκπαίδευσης. Εργάστηκα σε οργανώσεις νεολαίας, σε πολιτιστικές οργανώσεις Ασχολήθηκα και με το ποδόσφαιρο ε, και ρασιτεχνικά με την ηθοποία. Είχα αρκετά πλούσια πολιτική πείρα και ξεκάθαρες πολιτικές απόψεις. Αλλά αυτό είναι συνηθισμένο ε, για όλους τους πολιτικούς. Περιμένω να ισχύσουν οι δημοκρατικοί κανόνες και ως εκπρόσωπος μικρής περιοχής και χώρας θα ήθελα να εκλεγώ ω αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, γιατί θέλω να στρέψουμε την ε, προσοχή μα και στι μικρέ περιοχέ και χώρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τραβήξαμε κλήρο εδώ δύο ονόματα. Βαδίμ Τούντορ Κορνέλιου. Παρευρίσκεται ο κύριος Κορνέλιου. Ναι. Ναι. Απουσιάζει. Δώστε μου άλλο χαρτάκι. Έμα Μακλάκι. Ε, είστε εδώ. Ωραία. Άλλο ένα συνάδελφο να τραβήξω. Εμίλ Στογιάνοφ, τον είδα ναι, εδώ. ο κύριος Στογιάνοφ και η κυρία Μακλάρκιν. Παρακαλώ, ψηφολέκτες. Uh, uh, Ελάτε για την καταμέτρηση ε, των ψήφων στη συνέχεια. Λοιπόν, Έχουμε μία και μοναδική υποψηφιότητα, τον κύριο Σόινη. Μπορείτε στο ψηφοδέλτιο να γράψετε ναι, όχι ή το όνομα του υποψηφίου. Για και Σόινη σημαίνει ότι συμφωνείτε. Όχι σημαίνει ότι διαφωνείτε. Αν το ρίξετε λευκό, θεωρείται αποχή. Εντάξει, λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία. So, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σας συγχαρώ και εγώ μετά τους προηγούμενους συναδέλφους. Θα ήθελα να ζητήσω ε, να επαληθεύσουμε όπως και στις άλλες ε, επιτροπές, ότι οι αναπληρωτές έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν μαζί με τα τακτικά μέλη. Γιατί στι άλλε επιτροπέ, ε, στην πρώτη αυτή συνεδρία, σύσταση σε σώμα, είχαν το δικαίωμα ψήφου. Οι Αγαπητή κυρία Μωρέ, κοιτάξτε, στου συντονιστέ. Μόνο για την εκλογή των συντονιστών ισχύει αυτό που λέτε. Ψηφίζουν και τα τακτικά μέλη και τα αναπληρωματικά εξίσου. Για την Επιτροπή την ίδια ψηφίζουν μόνο τα πλήρη μέλη, τα τακτικά μέλη και αν κάποιος λείπει τον ε, αναπληρεί ένα αναπληρωματικό μέλο. Εντάξει. Λοιπόν, τα ονόματα. Λοιπόν. Μάτζε Κριστιάνο Άλαμ. Ελάτε να ψηφίσετε παρακαλώ. Α, δεν έχετε μοιράσει ακόμα τα χαρτιά. Καλά. Περιμένουμε. Yeah. Ναι. Έχετε πάρει όλοι ψηφοδέλτιο τώρα, όσοι δικαιούστε να ψηφίσετε εννοώ. Λοιπόν, αρχίζει η ψηφοφορία αλφαβητικά. Θα σας καλώ. Μάτζι Κριστιανό Άλαμ. Μαρία. Μαρία Μπατία Κουτσέτ. Please come here. Alam. Then Badia. Malika Benarab Atou. Lothar Biski. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Marie Honeyball. Sorin Katalin Ivan. Petra Kamerevert. Okay. Also, Madame Kammer-Ebert. Morten Lockegaard. Emma McClarkin. Marek-Henrik Migalski. Katarina Nevadolova. Frisula Pagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt. Ja, ja. Marco Scuria, Joanna Senissin. I apologize if it was. Timo Soini, Hannu Takula. Stojanov kommt später. Laszlo Tökesch.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 Ψηφίσατε όλοι, είχατε την ευκαιρία. Ωραία. Ολοκληρώνεται λοιπόν εδώ η ψηφοφορία και διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι οι ψηφολέκτες μας να καταμετρήσουν τις ψήφους. We can restart our meeting. Λοιπόν, επαναλαμβάνεται τη συνεδρίαση. Έχω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. If you are interested, you should listen. Αν σας ενδιαφέρει, ακούστε σας παρακαλώ πολύ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. So, 31... Λοιπόν, εψήφισαν 31 βουλευτές. 23 Τι αυτό. 23 ψήφοι είναι έγκυροι. Έγκυρες, Που σημαίνει ότι έχουμε λευκά άκυρα τα οποία δεν προσμετρώνται. 12 ήταν η πλειοψηφία που χρειαζόταν. 14 ψήφους πήρε κύριο Σουόνι ε, υπέρ και 9 όχι. Ε, εξελέγεται κύριε Σόνη. He has absolute majority. Έχει απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων και είναι σαφές ότι εξελέγει ο κύριος Σόνι. Παρακαλώ, ελάτε να καταλάβετε τη θέση σας. Now we go to the next. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο γύρο τώρα. So. Der Τρίτος αντιπρόεδρος. Παραμένει απαρτία. Δεν έχει φύγει κανονικά κανείς συνάδελφος από ό,τι είδα. Παρακαλώ κάντε τις προτάσεις σας για τον τρίτο αντιπρόεδρο. Παρακαλώ. Euh, Θα ήθελα και εγώ, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να σας συγχαρώ για την εκλογή σας, καθώς και τους υπολείπους αντιπροέδρους της Επιτροπής μας και εν ονόματι της Ευρωπαϊκή αριστερά τη ΓΚΟΕ να σας παρουσιάσω την υποψηφιότητα της ομάδας μας, του κύριου Λοτάρ Μπίσκι. Είναι ένας νέος ε, βουλευτής, αλλά επιπάντο από 15 χρόνια ήταν βουλευτής στην Bundesrat και Bundestag και ήταν και στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή ε, Πολιτιστικών Υποθέσεων της Γερμανικής Βουλής. Επί πολλά χρόνια ήταν πολύ διάσημος εκπαιδευτικός, δίδασκε για το κινηματογράφο και τα, και τα μέσα ε, ενημέρωση, για τα ΜΜΕ. Ευχαριστώ. Χάνου Τάκουλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, κύριο Σοίνη για την εκλογή του. Ελπίζω οι σοσιαλιστές να μην θελήσουν να γίνει και μια νέα ψηφοφορία. Νομίζω ότι είχαμε συμφωνήσει. Υπήρχε ένα πακέτο συμφωνίας. Εμείς θα υποστηρίξουμε τον κύριο Μπίσκι. Η Ευρώπη είναι πολυδιάστατη, πολύμορφη. Σεβόμαστε τις συμφωνίες που έχουμε συνάψει και ελπίζω και οι σοσιαλιστές στην Επιτροπή Πολιτισμού να σέβονται την πολιτιστική ποικιλομορφία της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Και εγώ δεν θεωρούσα ότι η Μαρία θα προτείνει τώρα κάτι τέτοιο. Παρακαλώ, Μαρία. Ευχαριστώ. Επειδή υπήρξε ένας προσωπικός υπενιγμός, εμείς ε, ανέκαθεν σεβόμαστε τον πλουραλισμό και την πολυφωνία. Και αν ζητήσαμε ψηφοφορία για τον προηγούμενο αντιπρόεδρο, δεν ήταν για προσωπικούς λόγους, γιατί δεν τον γνωρίζουμε προσωπικά τον κύριο Σόινι και είναι άξιος ε, σεβασμού. Απλώς η ομάδα στην οποία ανήκει είναι αντιευρωπαϊκή και δεν έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στις προτάσει τη ομάδα αυτή για την Ευρώπη. Γι' αυτό και κρατήσαμε θέση εποχής. Γιατί προσωπικά με τον κύριο Σουίνι δεν είχαμε τίποτα, κανένα πρόβλημα και θα συνεργαστούμε και με όλους τους αντιπρόεδρους αλλά και με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής όπως κάναμε ανέκαθαν. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Εάν δεν διαφωνεί κανείς με την υποψηφία του κυρίου Μπίσκη, παρακαλώ διαβοή να τον εκλέξουμε. Συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε, ελάτε να καταλάβετε τη θέση σας. Πάμε στον τέταρτο αντιπρόεδρο. Παραμένει η απαρτία. Äh, um Παρακαλώ, ποιος έχει να κάνει πρόταση. Χάνου, σήμερα τι έχεις την τιμητική σου, όλες οι προτείνεις. Κύριε που Ευχαριστώ, Ντόρις. Ναι, ξαναπέρα το λόγο. Χωρίς τους φιλελεύθερους δεν θα είχατε τέτοια ιδανική ομάδα, τέτοιο ιδανικό επιτελείο. Dream Team. Έχουμε τον κύριο Λούκερ Γκάρτ από τη Δανία να προτείνουμε μια σημαντική προσωπικότητα των μέσων μαζική ενημέρωση. Ευχαριστώ. Άλλε προτάσει υπάρχουν. Nicht der Fall zu sein. όχι από ό,τι φαίνεται. Παρακαλώ, συμφωνείτε. Und darf Lockegaard bitten, nach vorne zu kommen. Ελάτε παρακαλώ και εσείς στο Προεδρείο. Ich habe nicht gebeten, sich vorzustellen, nicht nötig. Ne? So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει ολοκληρωθεί το Προεδρείο. Θα ήθελα να σας ξαναπώ το εξή. Εκ δεξιών κάθονται οι άνθρωποι που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Εκτός από τους συμβούλους που έχουμε από τις πολιτικές ομάδες, επικεφαλής γραμματείας είναι ο ε, Στίβεν Τσόλτα ε, ε, και είναι ο κύριος Νάιταρ και η κυρία Kahn. ξεχνάω το όνομά της. Λοιπόν, οι τρεις εδώ της γραμματείας είναι εκείνοι που θα σας βοηθούν και όταν έχετε τις εκθέσεις σας, εκτός από τους συνεργάτες, τους προσωπικούς σας και των ομάδων, και βέβαια έχουμε και πάρα πολλούς ε, βοηθούς και γραμματείς και συνεργάτες πίσω, πολύ επιμελείς. Κάποια στιγμή θα συστηθούμε με ένα ποτήρι κρασί να γνωριστούμε και καλύτερα και πιο χαλαρά. Πάμε στο επόμενο θέμα τώρα της μέσης διάταξης που είναι ο προϋπολογισμός. Λυπάμαι πάρα πολύ που ήδη από σήμερα σας αναγκάζουμε να πάρετε απόφαση. Αλλά ε, στην περασμένη θητεία ήδη συζητήσαμε για τον προϋπολογισμό και θα πρέπει οπωσδήποτε το Σεπτέμβριο να έχουμε καταθέσει και ψηφίσει στην πρώτη ήδη ε, εβδομάδα συνεδριάσεων τις τροπολογίες μας για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου για φέτος. Λοιπόν, έχουμε την εξής κατάσταση. Πρώτον, χρειάζεται διορισμός εισηγητού ή εισηγήτριας τώρα για τον προϋπολογισμό εξ ονόματος Επιτροπής μας και επίσης να δούμε τι θα γίνει με τις τροπολογίες. Θα σας παρακαλούσα θερμότατα να ακολουθήσετε την εξής πρότασή μου. Τα τελευταία χρόνια είχαμε τη συνάδελφο και αντιπρόεδρο Χέλγα Τρούπελ, πολύ αξιόλογη που, ε, που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να την επιβεβαιώσουμε. Μέχρι τώρα έχει κάνει αυτή τη δουλειά και σήμερα θα ήταν πραγματικά άφρον να ορίσουμε άλλον εισηγητή που δεν έχει ιδέα και θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εξοικειωθεί με το θέμα αυτό. Εάν συμφωνείτε λοιπόν με την πρόταση αυτή και δεν διαφωνεί κανείς, τότε θεωρούμε ότι εξελέγει η κυρία Τρούπελ, επιβεβαιώθηκε η εισηγητρία. Ευχαριστώ. Ωραία καλείστε τώρα όλοι να ε, έχετε μελετήσει τον προϋπολογισμό, να μελετήσετε μάλλον τον προϋπολογισμό που θα λάβετε αύριο την Τρίτη, όπως έχει αυτή τη στιγμή και ποιες είναι οι αλλαγές που μπορείτε να κάνετε. Αύριο θα σας στείλουμε ηλεκτρονικά μία πρόταση. Παρακαλώ να τη μελετήσετε. Είναι η πρόταση του Συμβουλίου αυτή και εμείς μπορούμε ή έχουμε τη δυνατότητα να την τροποποιήσουμε. Αλλά υπάρχει προθεσμία για την κατάθεση αυτών των τροπολογιών που είναι η 31η Ιουλίου. 31η Ιουλίου. Μέχρι τότε θα πρέπει οπωσδήποτε αν θέλετε να κάνετε τροπολογία να την έχετε καταθέσει. Μπορείτε, γιατί είστε και μέλη της Επιτροπής και αναπληρωματικά έχετε τη δυνατότητα και το δικαίωμα να κάνετε τροπολογίες μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αν δεν το κάνετε δεν προλαβαίνει να μεταφραστεί, γιατί έχουμε τέτοιους περιορισμούς που έχουν να κάνουν με τις μεταφραστικές υπηρεσίες και τις χρονικές τους δυνατότητες. Αν θέλετε λοιπόν να κάνετε τροπολογία, αν σας πιέζει πάρα πολύ οπωσδήποτε και πρέπει να τη βγάλετε από πάνω σας, κάντε τη, αλλά αυτή τη βδομάδα ακόμα αν γίνεται για τη λίγη προθεσμία. Αν κάποιος θέλει να το μελετήσει, να το σκεφτεί καλύτερα για αργότερα, θα δούμε μέχρι ποια στιγμή μπορεί να κάνει τροπολογία, η οποία όμως θα μείνει αμετάφραστη. Πρέπει να την κάνετε στα αγγλικά ή στα γαλλικά από εκεί και πέρα, μετά τις 30 Ιουλίου. Εντάξει. Αυτή τη δεύτερη ημερομηνία δεν την γνωρίζουμε ακόμα, δεν την έχουμε ορίσει. Θα το κοιτάξει η γραμματεία μας και θα φροντίσει κάπου μέσα Αυγούστου να βρει μια τέτοια ημερομηνία, έτσι ώστε εκείνοι που θέλουν να πάνε διακοπές και να μελετήσουν τον προπολογισμό και τους κατέβηκα μια ιδέα μέχρι τότε, να μπορέσουν να την καταθέσουν. Πάντα στα πλαίσια των κονδυλίων που έχουμε, έτσι, στη διάθεσή μας. Λοιπόν, έχετε και αυτή την ευκαιρία επιπλέον. Από εκεί και πέρα όμως, μόνο στα αγγλικά ή στα γαλλικά, δεν απατώ, με επιτρέπετε επίση. Πάντω, εγώ θα σα συμβούλευα, ασχοληθείτε τούτη τη βδομάδα και αν οπωσδήποτε πρέπει να κάνετε τροπολογία μέχρι τι 31 Ιουλίου στη γλώσσα σα. Α, 12 το μεσημέρι, έτσι, 31 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Πέρας προθεσμίες για την κατάθεση των τροπολογιών. Τώρα, το Σεπτέμβριο έχουμε συνεδρίαση στις 2 και 3 του μηνός Σεπτεμβρίου. Και θα ασχοληθούμε με τη γνωμοδότηση αυτής της κυρίας Τρούπελ που θα την έχει εκπονήσει ως τότε για την πρόταση της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψε τότε 2 και 3 Σεπτεμβρίου και μετά μπορούμε στην πρόταση της κυρίας Τρούπελ να κάνουμε ξανά τροπολογίες μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν δύο δυνατότητες ακόμα να υποβάλουμε τις ιδέες μας και η ψηφοφορία για την πρόταση αυτή που λέγεται γνωμοδότηση της Επιτροπής και καταρτίζει η κυρία Τρούπελ και την καταθέτουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Αυτή η ψηφοφορία θα γίνει τον Οκτώβριο στη δική μας Επιτροπή για τη γνωμοδότηση. Τα είπα έτσι με αρκετή σαφήνεια. Τα εξήγησα καλά. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Η κυρία Τρούπελ μου διαβιβάζει ότι δέχεται να τη ανατεθεί ξανά η γνωμοδότηση και για τις περικοπές που έχει κάνει το Συμβούλιο στην πρώτη ανάγνωση, γιατί περί αυτού πρόκειται, σε τομείς που είναι της δικής μας αρμοδιότητας και σημαντική. Οι περικοπές λοιπόν αυτές του Συμβουλίου είναι κάτι που η ίδια θα ζητήσει να ακυρωθούν στη δική της νομοδότηση. Καλό θα ήταν λοιπόν να κάνετε τροπολογίες που να ανταποκρίνονται και να υποστηρίζουν τη δική της ε, πρόθεση. Έτσι. Να επανέλθουμε στο παλιό ποσό και όχι σε αυτό που έχει κόψει το Συμβούλιο. Αν έχετε τεχνικές ερωτήσεις, είναι στη διάθεσή σας πάντα η κυρία και η κυρία της Γραμματείας που σας είπα κάθονται εδώ δεξιά. Θέλει και η Κομισιόν να πει τίποτα, μήπω. Ποιο είναι εδώ, κύριο Νότσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πού είστε, εκεί πίσω, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Μπορείτε να συστηθείτε για να σας μάθουν και καινούργοι, παρακαλώ. Ε, Καλησπέρα. Είμαι τμήματάρχης στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό. Όπως είπε η κυρία Πακ, το Συμβούλιο, ο συνήθως, έχει κάνει διάφορες προτάσεις για να περιορίσει κάποιες δημοσιονομικές γραμμές σε σχέση με αυτό που είχε προτείνει η Κομισιόν. Να σας δώσω λίγο το πλαίσιο για αυτές τις περικοπές που έχουν προταθεί. Ε, κατατάσσονται σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα αφορά το πρόγραμμα που είναι συνεργασία με τις Ηνωμένε Πολιτείες και τον Καναδά. Δηλαδή συμφωνίες συνεργασίας με αυτές τις δύο χώρες ε, στον τομέα της εκπαίδευσης. Και τα τελευταία ένα-δύο χρόνια είχαμε προβλήματα εφαρμογής σε αυτά τα προγράμματα και σε αυτές τις γραμμές προϋπολογισμού. Όμως, ε, με την εκλογή του νέου Προέδρου στις ΗΠΑ φέτος, ε, παρατηρήσαμε μεγάλη πρόοδο στην εφαρμογή. Και υπάρχει πραγματικά μεγάλη θέληση για τη συνεργασία στι ΗΠΑ. Επίση, στον Καναδά ε, κάνουμε την ίδια παρατήρηση. Είχαμε προβλήματα, τώρα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ήδη από φέτο, στο βαθμό εφαρμογή, θα έχουμε πολύ καλύτερη κατάσταση. Υπάρχει μια συγχρηματοδότηση σε αυτή τη γραμμή του προπολογισμού και οι συνεργάτε μα, Καναδά και ΗΠΑ, συγχρηματοδοτούν κατά 50%. Η περικοπή που πρότεινε το Συμβούλιο τώρα, αν διατηρηθεί, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια νέα δυναμική, ή μάλλον η νέα δυναμική που υπήρχε σε αυτά τα προγράμματα θα καμφθεί. Τώρα, η δεύτερη γραμμή είναι μια παραδοσιακή γραμμή. Ε, το Συμβούλιο προβλέπει ε, περικοπή στα, δημο... στα διοικητικά έξοδα, στα προγράμματα εκπαίδευσης, ηθαγένειας και στο πρόγραμμα διαβίου μάθησης ε, για τα διοικητικά έξοδα περικοπή και το προπολογισμό που χρειάζεται η υπηρεσία για την εκτέλεση του προγράμματος υπό τον τίτλο 3β. Αυτή είναι μια κλασική περικοπή που ουσιαστικά την ακυρώνει η δική σας επιτροπή Έχουμε καλά επιχειρήματα για τις πιστώσεις πληρωμών. Έχουμε ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το τις, ε, τι πιστώσεις χρειαζόμαστε και για τις διοικητικές πιστώσεις. Έχουμε αυξήσει τις πιστώσεις αυτές ποσοστιαία, λιγότερο από τις δημοσιονομικές αυξήσεις που έχουμε προβλέψει. Επομένως, οι εκτιμήσεις μας είναι αρκετά ρεαλιστικές και δεν είναι καθόλου υπερβολικές και θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να ακυρώσετε αυτές τις περικοπές. Το τρίτο θέμα αφορά τις επισκέψεις μας, τα προγράμματα επίσκεψης. Είναι μικρά προγράμματα αυτά. Ε, λαμβάνουμε επισκέπτες από όλη την Ευρώπη, δεχόμαστε επισκέπτες από όλη την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια μικρή νέα πρωτοβουλία που θα θέλαμε να δοκιμάσουμε του χρόνου, επισκέψεις μαθητών από τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Θα θέλαμε να προωθήσουμε ε, κάποια πιλωτικά προγράμματα που μας κοστίσουν 300.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 300.000 ευρώ τα έχει κόψει το Συμβούλιο. Είναι ψυχία, αλλά πιστεύω ότι με αυτά τα λεφτά μπορούμε να κάνουμε κάτι χρήσιμο. Αυτά ήταν τα τρία θέματα τα οποία θα ήθελα να σας επισημάνω. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Is there any comment? Υπάρχει ένα σχόλιο από αυτόν που ακούσατε. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, βλέπω τις ε, δημοσιονομικές γραμμές και με νέο δεν καταλαβαίνω και πολύ καλά. Βλέπω ε, μία μειώση από 6 εκατομμύρια σε 1,5 εκατομμύριο. Ε, στον τίτλο για τον αθλητισμό. Προπαρασκευαστικέ δράσει στον τομέα του αθλητισμού. Αν κυρωθεί η θήκη τη Λισαβόνα, η δική μα επιτροπή θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τον αθλητισμό και μία πρόταση για περικοπή 85% του κονδυλίου για τον αθλητισμό. Τη στιγμή που η Λευκή Βίβλος και η συνθήκη της Λισαβόνας λέει ότι οφείλει να αφιερώσει κονδύλια στην προώθηση και την ανάπτυξη του αθλητισμού, είναι μια νόητη πρόταση, μια τέτοια κολοσσία περικοπή. Και μια τέτοια γνωστοποίηση της πρότασης ε, δυστυχώς θα έχει αρνητικές συνέπειες για το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Γιατί ο αθλητισμός ε, είναι πολύ σημαντικός για τους Ιρλανδούς και είναι ένας από τους ε, λίγους κλάδους που μπορούμε να προωθήσουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας έναντι της νίκης. Και νομίζω ότι μπορούμε να προωθήσουμε θέματα πολιτισμικά και αθλητισμού. Και με το σκεπτικό αυτό θα πρέπει να προτείνουμε αύξηση και σε καμία περίπτωση περικοπή και μάλιστα κατά 85%. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι. Δεν θα συζητήσουμε επί τη ουσία σήμερα για τον προλογισμό. Το Σεπτέμβριο θα το κάνω αυτό. Αλλά μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι η κυρία Τρούπελ ακριβώ αυτό θα κάνει που επιθυμείτε να ακυρώσει τι περικοπέ δηλαδή. Και έχετε δίκιο. Το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια ε, ζητάει να μπει ο αθλητισμός στις συνθήκες και εγώ ήμουν από τους πρωτοπόρους και αγωνίστηκα. Τώρα έγινε αυτό και το Συμβούλιο δεν το ήθελε ποτέ αυτό και έχει αρχίσει περικοπές. Ε, τώρα το αποφάσισε με το ζόρι περίπου, εμείς θα διταχθούμε σε αυτή τη ρύθμιση. Ο Ιβο Μπελέτ και ο Πάλι Σμιτ έχουν εργαστεί πάρα πολύ σε αυτά τα θέματα του αθλητισμού και εκεί θα βρείτε συμπαραστάτες και συναγωνιστές για να βοηθήσουμε τον αθλητισμό και οικονομικά τα επόμενα χρόνια. Και ερχόμαστε σε κάτι ακόμα που έχετε ε, στα χαρτιά σας για σήμερα που είναι το εξή. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν θα πρέπει να τα αφήσετε εδώ, να τα πάρετε μαζί σας. Είναι πολύ χρήσιμος ο οδηγός για νέα μέλη και για τους οδηγούς τους βοηθούς, συγγνώμη. Ένα οδηγό για τα νέα μέλη και του βοηθού. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη γραμματεία. Πρώτη φορά το κάνουμε. Είναι πολύ δύσκολη η αρχή για κάθε νέο και είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να δούμε πώ δουλεύει η Επιτροπή. Πολλέ φορέ είναι νέοι και οι υπάλληλοι, οι βοηθοί σα. Παρακαλώ πάρτε το μαζί και να το έχετε πάντα στο γραφείο σα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο οδηγό αυτό με πάρα πολύ πρακτικά στοιχεία πώ εργάζεται η Επιτροπή μα και ε, ένας κατάλογος πολύ χρήσιμων ε, ε, επαφών. Και κάτι ακόμα που έχετε στα έγγραφά σας, είναι το χρονοδιάγραμμα παρακαλώ, πάρτε το στα χέρια σας για το 2009. Το 2009, ναι. Το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων έχει ήδη αποφασιστεί, αλλά το αποφάσισε ακόμα αυτό το παλιό κοινοβούλιο και είχαμε την πρόνοια να αποφασίσουμε το χρονοδιαγράμμα μέχρι τα τέλη του έτους. Σα σας παρακαλούσα να κοιτάξετε τον κατάλογο αυτό και τις ημερομηνίες που απομένουν από το Σεπτέμβριο και μετά και να το δεχτείτε όπως έχει. Γιατί αν ανοίξουμε τώρα τους ασκούς του αιώλου, καήκαμε. Σας παρακαλώ, εντάξει φροντίσαμε να ε, εγκρίνουμε κάποιες ημερομηνίες. Παρακαλώ κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Μία παρατήρηση έχω μόνο για το χρονοδιάγραμμα. Αν, α, α, όπως προβλεφθεί, έχουμε την 9η Νοεμβρίου, συμπίπτει με την 20η επέτειο της κατάρρευσης του τείχου του Βερολίνου. Μία συμβολική ημέρα για πολλά έθνη και φαντάζομαι θα γίνουν πολλές διαδηλώσεις, οργανώσεις, εκδηλώσεις για τον εορτασμό αυτής επαιτίου, κάτι που θα εμποδίσει την παρουσία πολλών ευρωβουλευτών στη συνεδρίαση αυτή. Θα σας ζητούσα, θα, θα σας θέλω παρακαλούσα να μεταφέρουμε στην επόμενη και τη μεθεπόμενη ε, ή τη μεθεπόμενη μέρα την ημερομηνία της συνεδρίασης, γιατί η 9η Νοεμβρίου είναι πολύ σημαντική για όλη την Ευρώπη, να συνεδριάσουμε 10 ή 1 καταλάβω πολύ καλά και ιδιαίτερα ως Γερμανίδα αυτή την ένσταση. Αν δεν διαφωνεί κανένα άλλο να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την ημερομηνία. Προς τη 10η, 11η Νοεμβρίου θα προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω αν τα καταφέρουμε. Είναι και οι δυνατότητε που σας είπα και για τη μετάφραση και για τις αίθουσε. Τώρα ζητάει το λόγο ο κύριος Μπόρις και μετά ο κύριος Μάρτιν. E, Έχω μια πρόταση. Γιατί η 11η Νοεμβρίου είναι εθνική αργία στην ε, Πολωνία ε, και είναι η μέρα της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε Πολωνό μέλος στην ε, συνεδρίαση αυτή αν γίνει 11. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλο αργίες έχουμε. Αύριο είναι η σπουδότερη αργία του Βελγίου. Παρ' αυτά δουλεύουμε. Είναι η εθνική γιορτή στο Βέλγιο. 14 Ιουλίου δουλέψαμε στο Στρασβούργο. Τι άλλο έχουμε. 9 Νοεμβρίου φέτο είναι κάτι το ξεχωριστό και ιδιαίτερο. Είναι 20 ετία. Του χρόνου δεν θα το λάβουμε καν υπόψη μας. Θα προσπαθήσω. Έχω κατανόηση και για εσά, αλλά θα είστε και δικαιολογημένα από αν δεν έρθετε, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριο Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση ενημερωτικά που ίσως να μας ενδιαφέρει ε, τα νέα μέλη, εμείς που είμαστε νέα μέλη. υπάρχει καμία συνήθεια για το πότε συνεδριάζουμε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, ποια μέρα συνεδριάζει περίπου η Επιτροπή. Υπάρχουν συνήθειες τέτοιες για να ε, προγραμματίσουμε και το πρώτο εξάμεινο του 2010. Γιατί όσο πιο γρήγορα το προγραμματίσουμε νομίζω καλύτερο είναι αυτό. Υπάρχει τέτοια ρύθμιση. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε προτιμήσει εμείς εδώ σε ημέρες. Τώρα τυχαία στο δεύτερο εξάμεινο έχουμε τρεις φορές Δευτέρα Τρίτη. Την τελευταία φορά ήταν, ξέρω εγώ, Τρίτη ήταν να, τρει φορέ τρίτη. Δεν μπορώ να σα το πω εγώ αυτό τώρα. Αν επιθυμείτε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα ρυθμό να συνεδριάζουμε Δευτέρα και Τρίτη. Εάν θέλετε, ή Τετάρτη, Πέμπτη, ξέρω εγώ, όπως θέλετε. Πάντα περίπου τι ίδιε μέρες, Δευτέρα ή Τρίτη, για να προετοιμαζόμαστε καλά. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί ούτε ο πρόεδρο ούτε η Γραμματεία. Ξέρετε ότι είναι αλληλένδετο αυτό. Πολλές ε, επιτροπές συνεδριάζουν ταυτόχρονα και θα διαπιστώσετε αν είστε μέλη και σε άλλες επιτροπές, δεν θα έχετε πού να πρωτοπάτε. Εγώ θα προτιμούσα να έρχεστε πάντα εδώ βέβαια, αλλά αν είστε και μέλη αλλού και πρέπει να ψηφίσετε, βεβαίω θα πρέπει να πηγαίνετε εκεί και πάλι δικαιολογημένοι θα πόν Και εγώ θα το ζήσω αυτό, γι' αυτό άλλωστε έχω και τέσσερις αντιπροέδρους εδώ. Λοιπόν, το σημειώνω ως ε, ε, ε, παρότρινση, αλλά δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Η συνάδελφος από τη Γαλλία, παρακαλώ, κυρία Βερζιά. Ονομάζομαι Μαρία Κριστίν Βερζιά. Ήδη έχουμε συνεδριάσει και στις 14 Ιουλίου. 11 ε, Νοεμβρίου είναι ο ορτασμός ε, του, της λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου του, πολέμου, του πρώτου συγγνώμη, Παγκοσμίου Πολέμου που έγινε ένα από τα μεγαλύτερα μακελιά της ιστορίας. Νομίζω ότι ο εορτασμό ε, τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου είναι ιδιαίτερα σημαντικό γεγονό και συμβολικό. Μάλιστα. Ωραία. Είδαμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να ε, ε, αργούμε σε όλες τις εθνικές επαιτίους. Μπορούμε να τιμούμε και να έχουμε εκδηλώσεις, αλλά δεν μπορούμε να αλλάζουμε και να κυρώνουμε συνεδριάσεις επειδή έχει κάποιος γιορτή. Εδώ σα λέμε ότι είναι τα 20 χρόνια από την πτώση του τείχους. Πραγματικά ήταν αξιοσημείωτο γεγονό που πρέπει να το εορτάσουμε. Ε, άλλα θέματα μα κάνουν να είμαστε λυπημένου. να έχουμε μνημόσυνα. Αυτά με του πολέμου είναι μνημόσυνα. Μια γιορτή τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε για τα 20 χρόνια. Αν διαφωνείτε, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, μην κάνουμε τίποτα. Αλλά ε, βλέποντα τα πρόσωπά σα, είχα την αίσθηση ότι συμφωνείτε. Παρακαλώ. Um, also auf Deutsch. Να τα πω γερμανικά. Και βέβαια μπορεί κανείς να θεωρεί μια γιορτή πιο σημαντική από κάποια άλλη, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς όμως. Εγώ είμαι Πολωνή, άλλος έχει ζήσει τον κομμουνισμό, άλλος έχει ζήσει την Επανένωση, άλλος έχει ζήσει άλλες εθνικές γιορτές, την Επανάστασή του, ξέρω εγώ, τη 14η Ιουλίου. Για τους Γερμανούς η πτώση του τείχους είναι σημαντική και χαιρόμαστε που έπεσε, εν πάση περιπτώσει, αλλά θα πρέπει να διατηρούμε ένα ρυθμό κι εμείς εδώ. Και τώρα μπαίνουμε σε δύσκολη συζήτηση μην αρχίσουμε να συζητάμε πιανού οι γιορτές είναι σημαντικότερες τώρα. Ξέρω ότι για σένα είναι πρόκληση αυτό, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Μην ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, παρακαλώ. Πολύ συμβιλικό αυτό που μας είπες. Δεν το πρότεινα εγώ. Δεν ήταν δική μου η πρόταση. Μη Γερμανός, ε, να το πω έτσι, να το πω κι αυτό όμως. πριν συζητήσουμε για την 11η Νοεμβρίου, α κοιτάξουμε λίγο ότι στι 11 και 12 Νοεμβρίου έχουμε μία μήνυ ολομέλεια. Α κοιτάξουμε το χρονοδιάγραμμα δηλαδή του Κοινοβουλίου. Ούτω ή άλλω εκείνη τη μέρα δουλεύουμε. Μισή μέρα. Κοιτάξτε εδώ το χρονοδιάγραμμά σα παρακαλώ και δείτε την εργάσιμη για το Κοινοβούλιο. Μάλιστα, τελειώνει εδώ η συζήτηση. Δεν σα υπόσχομαι ότι θα αλλάξουμε την ημερομηνία θα το κοιτάξουν οι συντονιστές, στους οποίους εσείς εκλέγετε για να κάνω αυτές τις δουλειές, αν χρειαστεί. Ε, θα το ξανασυζητήσουν οι συντονιστές, θα δούμε αν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα. Αλλιώ, να μην αναλαθούμε σε αυτή τη συζήτηση τι είναι σημαντικό, τι δεν είναι. Όλα ε, σημαντικά είναι, αλλά ήταν θλιβερά, αλλά ήταν ευχάριστα. Σε όλα θα πρέπει να έχουμε ε, μνήμη και τιμή. Λοιπόν, επόμενη συνεδρία στη Δευτέρα και Τρίτη Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες που θα έρθει και ξεκούραστη μετά τις διακοπές με ιδέες για τον προϋπολογισμό. Σας εύχομαι καλές διακοπές, να ξεκουραστείτε από το στραπάτσο της προεκλογικής εκστρατείας και της αρχής εδώ που είναι πάντα χάος. Ευχαριστώ πολύ τους διερμηνείς για τη δουλειά τους και εμείς σας ευχαριστούμε και ελπίζω να μου διευκολύνετε τη ζωή τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, αριβεντέρτσι και χαίρετε. Γεια σας.